Uh, good morning, everybody. Um, welcome Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην σημερινή μας συνεδρίαση. Τα βασικά μας ζητήματα σήμερα είναι ότι να καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες σημαντικές ψηφοφορίες. Όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν ε, μαζί τους όλους τους υπευθύνους για τις ψηφοφορίες. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, καθότι μεταδίδεται η συνεδρία σε αυτή ζωντανά στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι παρακολουθούν τις ψηφοφορίες ζωντανά. Και να σας πω επίσης ότι έχουμε και ένα καινούριο ενημερωτικό φυλάδιο, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο και μπορείτε μάλιστα να εγγραφείτε στο διαδίκτυο στέλνοντας ένα email, να εγγραφείτε με συγχωρείτε σε αυτό το newsletter, το ενημερωτικό φυλάδιο. Λοιπόν, πολύ ο θόρυβος. παρακαλώ πολύ και προχωρήσουμε στις προφορίες. Να αυτό είναι το ενημερωτικό φυλάδιο. Αν θέλει κάποιος αντίγραφο υπάρχει. Στείλτε μας ένα email για να το λάβετε. Καλωσορίζω ιδιαίτερα κάποιους ε, προσκεκλημένους μας που ήρθαν στην ψηφοφορία τον πολύ καλό φίλο Βίτελ Μορέρα, τη Διεθνή Εμπορική Επιτροπή, από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αξίζει ένα χειροκρότημα. Από κοινού κάναμε πολλές καλές δουλειές και με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι 17 Μαρτίου θα γίνει ειδική ακρόαση εδώ για τις επιπτώσεις της ε, διατλαντικής εταιρικής σχέσης ε, στην ε, εσωτερική αγορά. Ελπίζω να είστε κι εσείς. Ευχαριστώ. Βεβαίως και θα είμαι. Και θέλω να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε και την Επιτροπή για την πρωτοβουλία και όλα αυτά που κάνετε για να αναβαθμιστεί το επίπεδο ενημέρωσης σε όλα αυτά τα θέματα. Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες τώρα. Έχετε τη σειρά. Θα αρχίσουμε με μια πολύ σημαντική έκθεση του εισηγητή Ανδρέα Σουάμπ για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή αν υπάρχουν κάποια θέματα και μετά θα αρχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να σας πω ότι ήταν πολύ ε, επικοδομητική η συνάντηση με όλους τους με τον Ραμόν, τους συναδέλφους από τους Πράσινους, τους Φιλελεύθερους, το ECR και με άλλες επιτροπές, ΛΥΜΠΕ, ΙΤΡΕ και μπορέσαμε να ε, καταρτήσουμε πολλές συμβιβαστικές και συμφωνούμε ότι στην ασφάλεια πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Ε, λυπάμαι που χρειάζεται να πάρω το λόγο τώρα, γιατί από νομική άποψη, δυστυχώ μόνο σε ένα θέμα, δεν είναι προσωπικό για μένα το θέμα, μου είπαν ότι πρέπει να είμαστε κατά τη προφορική τροπολογία, γιατί φαίνεται ότι ξεπερνά κατά πολύ το τι μπορεί να ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, ζητώ να μην το θέσετε σε ψηφοφορία. Λυπάμαι λίγο, γιατί συμφωνούμε ω προ το στόχο. Το ζήτημα όμω είναι ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητά μας. Αυτό είναι ο μόνος λόγος. Είναι η συμβιβαστική 27, η προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ όσους συμμετέσχουν στο φάκελο αυτό. Εντάξει, αρχίζουμε λοιπόν, γιατί ε, έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε αρκετά ικανοποιητικά. Ε, τροπολογία 138 Γκαρσές Ραμόν. Η κυρία Γκέπχαρτ σήμερα δίνει τον τόνο. Αρχίζουμε λοιπόν, ελέγχουμε και το ηλεκτρονικό σύστημα και θα δούμε και ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, τροπολογία 138. 34 μέλη. Όλοι έχουν τις κάρτες, όλα είναι εντάξει. Πηγαίνετε στο διπλάνο. «35 ψηφίσαντες πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 21 προς 11». Αφετ 16 υπέρ κατά δεκτή. Η 339 προσθήκη υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 140 του εισηγητή υπέρ. Παρακαλώ, υπέρ. Να δείχνετε σαφώς. Ευχαριστώ, κατά. Σαφώς δεκτή. Η 139 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 141 Ήτρε, αποκλειστική αρμοδιότητα, 142 του κυρίου Έγκστρομ υπέρ κατά αποχές δεκτή, 23 ως προσθήκη προσθέτομε fully respect υπέρ κατά απορρίπτεται, Ήτρε 40 υπέρ. Πρέπει να το ελέγξουμε αυτό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ήτρε 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφων. Ωραία. Απορριφθήκε λοιπόν. Ήταν 35 ψήφοι, 34 είπατε. Με τις 35, τις 35 ψήφους είμαστε εντάξει. Γιατί είχατε πει 34 κάποια στιγμή. Όχι, ε, είναι 35 οι ψήφοι. Ε, ενημερώνομαι εδώ από την οθόνη μου. Ψηφίζομαι το 143 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Λίμπε 48 υπέρ, κατά, δεκτή. Εκατόν μάντερς υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 41 τη ΣΥΤΡΕ, υπέρ, Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό. Ψηφίζουμε. Ήτρα 41 άρχεται η ψηφοφορία. Να ψηφίζετε αν γίνεται λίγο πιο γρήγορα παρακαλώ. Πατήστε γρήγορα το κουμπί. Πέρας. Λοιπόν, είναι ισοψηφία, απορρίπτεται λοιπόν με 16 υπέρ 16 κατά. Λίμπε 24. Πάλι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. I need you to vote more quickly, otherwise we'll be here all morning. Uh, it's lost. Ε, απορρίπτεται 15 υπέρ, 19 κατά. Να ψηφίζετε γρήγορα παρακαλώ. Άφετ 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 342 υπέρ κατά αποχές δεκτή ή 343 δεν θα την ψηφίσουμε 25 λίμπε υπέρ κατά απορρίπτεται ή 344 υπέρ κατά δεκτή 145 και άλλες ε, ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για να κάνουμε έναν έλεγχο. Την 146. Ψηφι... Υπέρ. Όχι, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, δεκτή. Δεκτή, δεκτή. 22. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ή 345 πίπτη. Λίμπε 27 ως προσθήκη. Υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 23 και 147 υπέρ. Κατά. Δεκτές. Θέλετε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτές. 25 προς 10. Ήτρε 46 αυτομάτως γίνεται δεκτή. Η 48 της Ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ταυτόσιμες τροπολογίες αυτές δεν θα τις ψηφίζουμε. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 21 υπέρ κατά δεκτή. Πάμε τώρα στην Ήτρε 50. Υπέρ. Ήτρε 50. Άρθρο 3, σημείο 8, β. Υπέρ. Νομίζω ότι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Όχι, την άφετη 20 νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα. Α, ναι, ναι, ναι, πήγα πολύ πιο κάτω. Αφετήκωση 20, ως προσθήκη, στην συμβιβαστική. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην Ήτρα 50. Υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι μάλλον γίνεται δεκτή. Α, δούμε, πέρας. Ναι. 19 υπέρ, 15 κατά δεκτή. Ήτρε 51 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ας το ελέγξουμε όμως, ας ελέγξουμε και αυτήν, γιατί είναι μικρή η διαφορά. Ήτρε 51, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίφθη. Απερίφθη. Καλά που το ελέγξαμε. 26 και ήτρε 52. Μαζί με την 27 και 53. Τέσσερις μαζί Πέρ. Κατά δεκτές σαφώς. Οπότε τώρα πάμε στην Ήτρε 54, έτσι δεν είναι. Ήτρε 54, Επιτροπή Βιομηχανίας. Πέρ. Ε, ήταν μέρος του, της ομάδας. Α, όχι, όχι, όχι, ήταν μαζί με τις άλλες. Πάμε στο άρθρο 4, 152, δηλαδή να διαγραφεί όλο το άρθρο υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οπότε οι επόμενες δύο καταπίπτουν. 154 συνδέεται με τη συμβιβαστική 6, οπότε πάμε στην 155 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, Ήτρε 56, τμηματική ψηφοφορία, πρώτο μέρος ε, της 56, περ, κατά, αποχές, ε, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Ή 156 και Ήτρε 57, υπέρ, υπέρ, κατά, δεκτές αφώς Η Λίμπε 29, καταπίπτει η 157 του κυρίου Έγκστρομ είναι προσθήκη όμως υπέρ έλεγχος ως προσθήκη 157 άρχεται η ψηφοφορία λίγο πιο γρήγορα παρακαλώ πέρας απερίφθη αυτή 18 προς 15. Κάποιος έφυγε, είναι 34 οι ψηφίσαντες. Τώρα, τροπολογία 30 και ήτρε 58 υπέρ. Κατά δεκτές 158 υπέρ. Κα... όχι, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά να δούμε. Πέρας. Ναι. Απερίφθη. 159 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 160 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 161 του κυρίου Έγκστρομ υπέρ. Κατά. Δεκτή. Λίμπε 30 ως προσθήκη υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Λίμπε 31 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 31 και 59 υπέρ, κατά, δεκτές, ε, αποσύρθηκε 32. Η 162 του εισηγητή υπέρ, κατά, σαφώς ναι, 60 ε, καταπίπτει, 33 και άφετ 21 υπέρ. Κατά. Α, καταπίπτει. Α, ναι, ναι, ναι, καταπίπτουν γιατί η 162 έγινε δεκτή. Πάμε στην 163 του κυρίου Γκαρσές Ραμών. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 164 και 61 ε, μαζί με την 34, 36 υπέρ. Κατά δεκτές όλες αυτές. Οπότε τώρα πάμε στην 165 του εισηγητή υπέρ. Κατά δεκτή 166 υπέρ. Κατά δεκτή 38 και ήτρα 67 υπέρ. Κατά δεκτές Λίμπετρι ε, καταπίπτει 66 ήτρε ως προσθήκη υπέρ κατά για να το ξαναδούμε ποιοι είναι υπέρ όχι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ήτρε 66 ως προσθήκη άρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη με διαφορά μιας ψήφου Λίμπε 35 υπέρ κατά απορρίπτεται 39 και 68 υπέρ κατά δεκτές Ήτρα 69 όλα αυτά αυτομάτως γίνονται δεκτά πάμε στη συμβιβαστική 22 ε, ψηφίζουμε είναι τμηματική ψηφοφορία που τη ζήτησε η Άλντε ε, πρώτο μέρος της 22 υπέρ κατά δεκτό και το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 22 υπέρ κατά δεκτό. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 23 υπέρ κατά δεκτό. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά δεκτό. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά δεκτή και έτσι πάμε στην 192 του κυρίου Έγκστρομ υπέρ κατά απορρίπτεται 193 υπέρ κατά απορρίπτεται 53 και 80 υπέρ κατά δεκτές λίμπε 40 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρε 81 υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ήτρε 81 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με διαφορά μιας ψήφου. Συμβιβαστική τροπολογία 26 υπέρ. Κατά δεκτή Ήτρα 82. Υπέρ. Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ήτρα 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 31 ε, ψήφισαν. Πού είναι οι άλλοι. Απορρίφθηκε όμως. 31 ψήφισαν. Ε, είναι 34 οι κάρτες. Έχει απορριφθεί πάντως με σαφή διαφορά. Συμβιβαστική 27 χωρίς την ε, προφορική τροπολογία. Στις προφορικές υπέρ, κατά δεκτό. Πάμε τώρα. Άφετ 26 υπέρ, δηλαδή κατά δεκτή. Α, ξανά, όχι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άφετ 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε άφετ 27 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε 197 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 198 ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οπότε πάμε στη συμβιβαστική 29 υπέρ κατά δεκτή και πάμε τώρα στη συμβαστική 30 υπέρ κατά δεκτή συμβιβαστική 31 υπέρ κατά δεκτή 226 ως προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται ήτρε 90 όχι Πάμε στην άφετη 28 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Άφετη 29 υπέρ. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την άφετη 29, άρχεται η ψηφοφορία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων νομίζω απορρίφθηκε αλλά να το βεβαιώσουμε. Όντως απερίφθη. Μπλοκ, το επόμενο δεν ψηφίζεται. Πάμε στην συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά δεκτή. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 228 προσθήκη. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Πάμε τώρα σε αιτιολογικές, ε, τις αναφορικές προτάσεις, 106 τροπολογία υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Την 106. Δεκτή με διαφορά δύο ψήφων. 107 ε, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Άφετ 1 υπέρ κατά απορρίπτεται. ΛΥΜΠΕ 1 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρα 1 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά δεκτή. Άφετ 3 υπέρ κατά απορρίπτεται. Άφετ 4 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 111 υπέρ κατά απορρίπτεται. Άφετ 6 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 4 τμηματική ψηφοφορία. Το ζητούν οι πράσινοι. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ, κατά δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά και αυτό δεκτό. Τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ, κατά δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά δεκτή. Ήτρε 5 υπέρ, κατά δεκτή. Ήτρε 6 υπέρ, Άρχεται η ψηφοφορία στην 6. Ήτρα 6 ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. Άφεται 9. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 112. Δεν θα ψηφίσουμε αυτήν. 113 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά δεκτή. Λίμπε 5 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά δεκτή. 115 υπέρ κατά δεκτή. Λίμπε 6 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Άφετ 10 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρε 9 υπέρ κατά δεκτή. Λίμπε 7 ως προσθήκη υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά δεκτή. Ήτρε 12 υπέρ κατά δεκτή. Άφετ 11 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά δεκτή. Ήτρα 14 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά δεκτή. 9 ε, της Λίμπε υπέρ κατά απορρίπτεται. Ε, Ήτρα 17 υπέρ κατά δεκτή. Η λίμπε 10 καταπίπτει, λίμπε 11 υπέρ, κατά απορρίπτεται, συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά δεκτή, 122 υπέρ, κατά απορρίπτεται, ήτρε 19 υπέρ, κατά απορρίπτεται, ήτρε 20 υπέρ, κατά δεκτή ε, τροπολογία 7 και ήτρα 21 υπέρ κατά αυτοί, αυτές γίνονται δεκτές συμβιβαστική 13 υπέρ κατά δεκτή λίμπε 13 υπέρ κατά απορρίπτεται 124 καταπίπτει συμβιβαστική 14 Λάθος έκανα. Ε, θα ψηφίσουμε την 124. Θα την ψηφίσουμε ε, από μόνη της, όχι προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Δεκτή, κύριε Έγκστρομ, συγγνώμη. Συγγνώμη που πήγα να σας αποκλείσω. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Λίμπε 15. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρα 25 υπέρ κατά απορρίπτεται 12 υπέρ κατά δεκτή λίμπε 16 υπέρ κατά απορρίπτεται 125 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 περ κατά δεκτή. Τροπολογία 126 ως προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά δεκτή. Η Λίμπε 18 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά δεκτή. Ε, άφετ 13 υπέρ κατά απορρίπτεται. Λίμπε 19 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 130 υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 130. απορρίπτεται 15 υπέρ 19 κατά. 131 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά δεκτή. Ήτρε 30 υπέρ κατά δεκτή. Άφετ 14 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρε 31 υπέρ κατά δεκτή. Λίμπε 20 ως προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται. Πάμε στην 133 με την προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ. Κατά δεκτή. Αφ, όχι. Ε, ήτρε 32 υπέρ. Ναι, ήτρε 32 υπέρ κατά δεκτή. Άφετ 15 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρε 33 υπέρ κατά απορρίπτεται. Δεν την ψηφίζουμε τη 18. 134 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά δεκτή. Ήτρε 34 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 135 με την προφορική υπέρ κατά δεκτή. Ήτρε 35 ως προσθήκη υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 20 και 37 της Ήτρε υπέρ κατά δεκτές. Λίμπε 21 προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 21 και ήτρα 38 υπέρ, υπέρ, κατά, δεκτές. Και λίμπε 22, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε όλο το σχέδιο έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με 33 υπέρ, με μία ψήφο κατά και μία αποχή. Δίνω το λόγο στον εισηγητή για να μας πει για την διαπραγματευτική εντολή. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ψήφισαν θετικά. Πρέπει σύντομα να θυμηθούμε ότι είναι κρίσιμο το θέμα, όμως βρήκαμε συμβιβαστική λύση μεταξύ σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων. Μπορεί καμιά φορά οι διαφορές να είναι μεγάλες σε θέματα τεχνολογίας, ε, ε, της πληροφορίας, αλλά βρίσκουμε λύση. Ευχαριστώ όλους. Ελπίζω να αρχίσουμε με άτυπες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πραγματικό τριμερή διάλογο, αλλά αν κινηθεί γρήγορα το Συμβούλιο μπορεί και αυτό να γίνει. Ε, θα ήταν πολύ καλό να μου δίνετε αυτή την εξουσιοδότηση, αυτή την εντολή. Ναι. Θα ψηφίσουμε και γι' αυτό ηλεκτρονικά για να δώσουμε εντολή στον εισηγητή να αρχίσει άτυπες συζητήσεις με το Συμβούλιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι. Γιατί βλέπω 32 ψήφους, πάντως είναι αρκετές νομίζω. Πέρας. Σαφής εντολή που ελάβατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, Ανδρέα Σβάμπ και όλους τους σκιώδης και τους συντάκτες νομοδοτήσεων. Πολύ καλή δουλειά. Επόμενο θέμα. Έκθεση του κυρίου Μάντερς απλούστευση της μεταφοράς ε, μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο εισηγητής θέλει να μιλήσει. Να σας πω μόνο ότι ξεκινήσαμε ατύπως ε, τον τριμερή διάλογο και τουλάχιστον βλέπουμε ότι υπάρχει μια κάποια συνεργασία με το Συμβούλιο. Ενδεχομένως λοιπόν την Δευτέρα η ομάδα εργασία Συμβουλίου να καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Μπορούμε πάντως να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για το σημαντικό αυτό ζήτημα και ενδεχομένω να καταφέρουμε να πετύχουμε συμβασμούς για τα μεγάλα ζητήματα. Και αν πετύχουμε για τα μεγάλα, ενδεχομένω να πετύχουμε συμβασμούς και για τα μικρότερα ζητήματα. Θέλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή όμως ε, και ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να δώσουμε στον κύριο Μάντερς και στους κοιόδη εισηγητές μία εντολή διαπραγμάτευσης. Άρχεται λοιπόν ψηφοφορία για την εντολή αυτή τη διαπραγματευτική. Πέρας. Ξεκάθαρα λοιπόν η εντολή που σας δίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ πέρα, παρακολουθεί τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλει ο εκπρόσωπος Επιτροπής να πει κάτι. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που δόθηκε εντολή στον εισηγητή σας. Πολύ ωραία, ο Πρόεδρος. Θα δούμε πώς θα προοδεύσουμε για το ζήτημα αυτό. Περνάμε στο επόμενο σημείο, την επόμενη ψηφοφορία όπου χρειάζεται να εγκρίνουμε επισήμως τα συμπεράσματα για την διαθεσιμότητα ράδιο εξοπλισμού στην αγορά, τα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων. Η κυρία Βάλια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε προχωρήσει λίγο παραπέρα από τον κύριο Μάντερ, στον οποίο εύχομαι καλή επιτυχία με τη νέα Προεδρία. Είχαμε τα βασικά, τα είχαμε κάνει επί Λιθουανικής Προεδρίας και τώρα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες, διότι αν δεν είχαμε από κοινού πραγματικά ε, δώσει μάχη για τη θέση της Επιτροπής, δεν θα είχαμε τελειώσει σήμερα, διότι το Συμβούλιο δεν βοήθησε πάντοτε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους λοιπόν και τους συνεργάτες μας και την κυρία Φαλάισερ ήταν πολύ θετική συνεργασία, ευχάριστη με τους συναδέλφους και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Ε, well, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχω την επίσημη επιστολή από το Συμβούλιο με το σχετικό κείμενο. Πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε το κείμενο αυτό. Άρχεται ηλεκτρονικός ψηφοφορία. Άρχη ψηφοφορία για την έγκριση των ε, συμπερασμάτων των διαπραγματεύσεων για τη διαθεσιμότητα στην αγορά. Νομίζω ότι πραγματικά έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ στο να βελτιωθεί η οδηγία πέρας, λοιπόν, και σαφώς λοιπόν εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ, δύο κατά. Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την κυρία Βάιλερ, η οποία ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν ε, σαφές το αποτέλεσμα στο παρελθόν, δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν. Ξέρετε ότι οι τεχνικές αυτές οδηγίες πολλές φορές κρύβουν και διάφορες εκπλήξεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, όπου θέλουμε να εγκρίνουμε επισήμως Επίσημη έγκριση προφορικής ερώτησης για την αξιολόγηση εθνικών καονιστικών ρυθμίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα επαγγέλματα. Εργαστήκαμε πάρα πολύ όλε οι πολιτικέ ομάδε για το ζήτημα αυτό. Πρέπει να εγκρίνουμε το ζήτημα αυτό επισήμω. Την προφορική δηλαδή αυτή ερώτηση. Άρχεται η ψηφοφορία για την έγκριση προφορική ερώτηση. εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Θα συνεργαστούμε λοιπόν προκειμένου να καταφέρουμε να εντάξουμε την προφορική αυτή ερώτηση στη μέρη διάταξη της Ολομέλειας πολύ σύντομα. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Λόκεγκάρτ, ιδίας πρωτοβουλίας όσον αφορά το Solvit. Κύριε Λόκεγκάρτ, κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, προφανώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές. Θεωρώ ότι είχαμε μία καταπληκτική συνεργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι στα πλαίσια της Επιτροπής μας έχουμε μία ευρεία συνένεση για το ζήτημα αυτό. Κατάφερα λοιπόν, καταφέραμε λοιπόν από κοινού να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα τόσο προς την Κομισιόν όσο και προς τα κράτη-μέλη προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το προτινόμενο εδώ σύστημα. Ξέρετε ότι το ζήτημα του Solvit θα μας απασχολήσει βέβαια και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία για όσου από εμά παραμείνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα ευθύ αμέσω με την ψηφοφορία. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Απασχόλης 5, καλύπτεται από τη 12, 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 ως προσθήκη 13 με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Έμπλ 1 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 15, ψηφίζουμε την τροπολογία 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 16 καταπίπτει. Περνάμε στη βασική τροπολογία παριθμών 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10. 18 ως προσθήκη στην παράγραφο 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έμπλα 7 καλύπτεται. 21 υπέρ κατά, εγκρίνεται. 22 προσθήκη, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οι 28-29 καταπίπτουν, περνάμε στην έμπλη 3, η οποία καλύπτεται από άλλη, 30 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 30. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφι υπέρ, 13 κατά, 31 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Έμπλ 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 32 καταπίπτει και η 34 επίση Employment 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. 21, μάλλον 35 διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 35 για την παράγραφο 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 36 καταπίπτει, 37 επίσης, 38 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 40 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 41 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, συμβασική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 47 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 48 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 49 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθμών είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται, 2 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 3 υπέρ, κατά εγκρίνεται, τροπολογία 4 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 5 υπέρ, κατά γκρίνεται, Έξι, υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρτη ψηφοφορία για την τελική έκθεση. Πέρας. Εγκρίνεται 33 ψήφοι υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λόκεγκάρτε. Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε λοιπόν στη μερίστη τη Ολομέλεια και την έκθεση αυτή του στο μότερο δυνατό. Περνάμε τώρα στη δική μου την έκθεση. Α ψηφίσουμε λοιπόν την δική μου την έκθεση. Ο κύριο Φόξ αποχωρεί. Λοιπόν, α ψηφίσουμε τη δική μου την έκθεση παρακαλώ πολύ. Δείξτε λίγη υπομονή. Ξέρετε ότι είναι πολύπλοκος ο κατάλογος ψηφοφοριών γιατί χρειάζεται και να γίνει μία αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση κάπως της έκθεσης αυτής. Υπάρχουν αρκετές συμβαστικές τροπολογίες καθώς επίσης και αρκετές κατά τμήματα ψηφοφορίες. Να ευχαριστήσω πάντως τους κοιόδης συγητές για την επικοδομητική τους συνεργασία. Σας πενθυμίζω ότι πρόκειται για μια γνωμοδότηση η οποία υποβάλλεται προς την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ψηφίσουμε όμως για τμήματα τα οποία έχουν να με τους καταναλωτές που είναι ουσιαστικά δική μας αρμοδιότητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 98 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κα... Άρχεται μάλλον ψηφοφορία για τροπολογία 101. Πέρας εγκρίνεται 19 προς 16. 102 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ κατά απορρίπτεται. 104 και 105 από κοινού υπέρ κατά εγκρίνονται. 106 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ κατά απορρίπτεται. Αποσύρεται 108, η 109 έχει εγκριθεί αυτομάτως, 110 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 11 ως προσθήκη, μάλλον η 111 πρώτα, τροπολογία 111 ως προσθήκη υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον για την τροπολογία 111 ως προσθήκη. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με διαφορά μιας ψήφου. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 116 του κύριου Έγκστρομ υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11 με χωριστή ψηφοφορία. Βλέπετε τα δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της συμβαστικής 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 122 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 135, 136, 137 και 138 μαζί υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 140 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 143 και 144 ταυτόσιμες υπέρ κατά απορρίπτονται. 145 υπέρ κατά απορρίπτεται 146 υπέρ κατά απορρίπτεται 147, 148, 149 πρόκειται για διαγραφή και τρεις μαζί υπέρ κατά απορρίπτονται 150 α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος εγκρίνονται. Εγκρίνεται λοιπόν η προτινόμενη διαγραφή. Περνάμε στην... Τροπολογία 5, λέει ο Πρόεδρος, για το άρθρο 22, τροπολογία 5, για να καταλάβετε ακριβώς τώρα τι ψηφίζουμε. Θα θυμάστε ότι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε από κανονισμό σε οδηγία. Έπρεπε να γίνουν λοιπόν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές. Έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε όλες τις τροπολογίες ώστε να συνάδουν με μια οδηγία. Υπέρ λοιπόν της 5, κατά, εγκρίνεται. αν μάλλον μπορούμε να προχωρήσουμε στην 158 λέει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική τροπολογία 12, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική τροπολογία 13, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 186, 187 μαζί υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 188 και 189 έχουν εγκριθεί. Πάμε στην βαστική 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 192 και 209 μαζί υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 από τον εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Την έχουμε καλύψει μάλλον, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε στην 284, λίγες σελίδες πιο κάτω. Περνάμε δηλαδή στη σελίδα 16 και ψηφίζουμε την τροπολογία 284 της κυρίας Μπάστος. Με παρακολουθείτε υπέρ, κατά εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 254 προσθήκη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 3, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Έχουμε ισοψηφία. Περνάμε Στην 23 υπέρ κατά εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 270 προσθήκη υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 309 του κύριου Κρόιτσμαν. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οι 33 και 310 καταπίπτουν. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 39 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 40, η 41, 43 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 325, 326 υπέρ κατά εγκρίνονται. 327 υπέρ κατά Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 327 παρακαλώ. πέρας, εγκρίνεται. Οι 329 και 330 από κοινού, υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Οι 328 καταπίπτει, η 331 τώρα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 334 υπέρ, με συγχωρείτε, διακόπτει ο πρόεδρος, 333 μάλλον, υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 334 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 335 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 336 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, τροπολογία 338 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 340, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 342 φορά διαγραφή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 343 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 344 υπέρ, Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 344, άρτη ψηφοφορία. 35 οι ψηφίσαντες, πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά δύο ψήφων. Εγκρίνεται λοιπόν και περνάμε στην 46. Τροπολογία 46. Υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 46 ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 16 κατά. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 53 και 54 μαζί υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 55. 56 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 59 υπέρ κατά εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 60, 61 και 62 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται. Η 63 απορρίπτεται αυτομάτως και ψηφίζουμε την 64 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 65. Δεν την ψηφίζουμε, μάλλον 66 υπέρ κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 69 και 70 δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε. Τι κάνουμε τώρα με την 71. Ψηφίζουμε τροπολογία 71 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 72 κατά πίπτη, 73 δεν ψηφίζουμε, 74 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 77 και 78 έχουν εγκριθεί. 80 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 81 καταπίπτει, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε την 79 προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Πράγμα που σημαίνει ότι 83 και 84 καταπίπτουν. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ. ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 87. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 89. Τι κάνουμε τώρα με την 90 και 91. Περνάμε στην τροπολογία 93 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 95. Μάλλον 96 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95 καταπίπτει. Τροπολογία 97 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης και θα ήθελα την υποστήριξή σας προφανώς προκειμένου να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 35 ψήφοι περ μία κατά και καμία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας και θα διαπραγματευτώ λοιπόν περισσότερο με την Επιτροπή Βιομηχανίας για το ζήτημα αυτό. Good. Πάμε στην τελική μας, τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. Για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2014, του Αντιπροέδρου μας κυρίου Κοφεράτη, μήπως θέλετε να πείτε τίποτα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές για την διαθεσιμότητά τους, καθώς επίσης και το προσωπικό τους, τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μας βοήθησαν να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και να φέρουμε εις πέρα στην έκθεση αυτή, η οποία τελικά ήταν πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι φαινόταν στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Τροπολογία 6, παράγραφος 1, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. 7, ε, συγγνώμη, υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 10 υπέρ. Κατά. Α, υπέρ. Κατά. Οι φιλελεύθεροι ψηφίζουν καθόλου. Μιλάω για την τροπολογία 10. Και δική μου. Παρακαλώ να ψηφίσετε λοιπόν. Είναι καλή τροπολογία. Ωραία. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 57 Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά εγκρίνεται. 33-34 καταπίπτουν. 35 υπέρ κατά εγκρίνεται. 36 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά απορρίπτεται 62 υπέρ κατά εγκρίνεται 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εγκρίνεται 63 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 41, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 46, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά α, α, εγκρίνεται 50 υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε σε αιτιολογικές σκέψεις 1 υπέρ κατά εγκρίνεται 2 υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 4 υπέρ κατά εγκρίνεται και 5 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την ε, τελική γνωμοδότηση. Την τελική έκθεση, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, κύριε εισηγητά. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικός. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 34 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια κύριε Κοφεράτη. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ψηφοφορία αυτή. Τελειώσαμε πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Ξέρω ότι ο κύριος Μπίλαν έχει προετοιμάσει μία σημαντική έκθεση για να τη συζητήσουμε, όμως νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εδώ. Θέλετε να περιμένουμε λιγάκι, γιατί πρέπει να έρθει και η Επιτροπή. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, περίπου 10 λεπτά. Γιατί οι κύριοι Μπίλαν μας ενημέρωσαν ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταφθάνουν. Μπόρισοφ, Βερνιό είναι εδώ ως σκιώδης, ως σκιώδης εισηγητές για τους φιλελεύθερους θα πρέπει να είναι εδώ ο κύριο Σμιτ. Τον κύριο Ντε δεν τον βλέπω. Λοιπόν, 10 λεπτά διακοπή, οπότε 11 παρά 20 ξαναρχίζουμε. Έχετε χρόνο για ένα καφεδάκι. Μιλάμε για τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξη πληρωμών με χρήση καρτών, όταν επανέλθουμε στις 11 παρα 20. Ο κύριος Μπορίσοφ είναι εδώ, η κυρία Βερνιό είναι εδώ ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, που είναι σκιώδης εισηγήτρια για τους ε, σοσιαλιστές. Είναι σημαντική αυτή η γνωμοδότηση, γιατί είναι πραγματικά ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα θα συζητήσουμε τις 91 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, αλλά περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί, όπως είπα, τελειώσαμε νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ για την αποτελεσματικότητά σας. Right. Well, thank you um, uh, for uh, uh, assembling again after the votes. Um, I'm very grateful. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε. Συγγνώμη που ε, βιαστήκατε να έρθετε. Τελειώσαμε λίγο νωρίτερα τις ψηφοφορίες. Την, την επόμενη φορά θα σας ειδοποιήσουμε νωρίτερα. Νομίζω η κυρία Βέιζεμπεκ είναι εδώ. Έχει ξαναέρθει στην Επιτροπή μας. Ε, περιμένουμε κανέναν άλλον από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚΤ. Θέλετε να αρχίσουμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δουλεύουμε τώρα για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση των, ε, της Επιτροπής ΕΚΟΝ για μια πρόταση για κανονισμό διατραπεζικών προμηθειών ε, για πράξη πληρωμών με τη χρήση καρτών. Ήταν, ε, είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό είναι πολύ σημαντική η πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει σημαντικές συνέπειες για τους καταναλωτές. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερη σημασία ε, για την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Ο Άνταμ Μπίλαν είναι ο εισηγητής μας, έχουμε τον κύριο Μπόρισοφ, ε, έχουμε την κυρία Βερνιό, νομίζω ότι ο κύριος Μάντερς έρχεται και εκείνος για να εκπροσωπήσει τον κύριο Σμιτ. Δεν νομίζω ότι οι πράσινοι έχουν ε, σκιώδη εισηγητή, αν θυμάμαι καλά, και ελπίζω ότι και οι φιλελεύθεροι θα έρθουν. Λοιπόν, να αρχίσουμε τότε, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπίλαν, για να μας πει ποια είναι η άποψή του για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί ως τώρα. Εκτός από τις δικές σας 19 ε, τροπολογίες, ε, εσείς λάβατε άλλες 80. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε την αναβολή για σήμερα του θέματός μου. Δεν μπορούσα να είμαι εδώ εχθές. Και επειδή είναι αρκετά λεπτομερείς οι σημειώσεις μου, θα μιλήσω πολωνικά. dotyczące interchange e, wywołuje dużo emocji i jest przedmiotem είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και υπήρξε... Υπήρξαν ε, πολλές τροπολογίες, ε, οι οποίες πολλές περιπτώσεις αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από αυτά που είχα συμπεριλάβει εγώ στη γνωμοδότησή μου. Υπάρχουν τροπολογίες τις οποίες βλέπω τη δυνατότητα συμβιβαστικών τροπολογιών και μιλάω για, την τροπολο... για τις τροπολογίες που αφορούν τους ορισμούς των ε, πληρωμών με χρήση καρτών ε, και χρεωστικών καρτών, ε, της τροπολογίας του κυρίου Ντεγιόν και τις δικές μου τροπολογίες 36 με 39. Το ίδιο ισχύει και τις τροπολογίες για τον ορισμό της, των πιστοτικών καρτών. μιλάω για την τροπολογία 9, όπως επίσης και για τη μεταβατική περίοδο στα άρθρα 3 και 4, δηλαδή τροπολογίες 62, 60, 62, 64 και 65 και τις δικές μου τροπολογίες 14 ε, και 15. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά τα σημεία υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ε, συμβαστικών τροπολογιών. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο των προμηθειών, ε, των τελών, Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με, την, με το σταθμισμένο όρο και θα επανέλθω σε αυτό για τις ε, τροπολογίες της κυρίας Βερνιό. Ε, τις γνωρίζω, ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένα κράτη-μέλη που προσαρμόζονται στις προτινόμενες διατάξεις. Δεν ε, έλαβα υπόψη, δεν ε, σκέφτηκα εγώ ένα ενιαίο τέλος, αλλά είμαι ανοιχτός σε αυτό. Ίσως στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών στο Στρασβούργο να φτάσουμε σε συμφωνία για το θέμα αυτό. Επίσης, συμφωνώ με την τροπολογία 79, 87 και 70. Ε, μου αρέσουν αυτές οι τροπολογίες. Να συνεχίσω τώρα σε ορισμένα από τα σημαντικά ε, ζητήματα τα χαμηλότερα τέλη σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στο κανονισμό. 54 και 68 Στήλερ και 69 Μπορίσοφ. Για αυτές τις τροπολογίες μιλάω. Δεν βλέπω σοβαρά προβλήματα με αυτές τις τροπολογίες, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρω αν χρειάζονται ε, αν είναι απαραίτητε, γιατί το ή τα κράτη-μέλη ε, έχουν τη δυνατότητα να έχουν χαμηλότερα τέλη. Αν δείτε για παράδειγμα το 18 των αιτιολογικών αναφορών, λέει ότι ο κανονισμός δεν πρέπει να απαγορεύει στα κράτη-μέλη να έχουν χαμηλότερα ανώτατα όρια ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για να επιτύχουν τον ίδιο σκοπό. Το επόμενο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι για τις παραγράφους 1, 2, άρθρα 3 και 4. 53 και 67 τροπολογίες της κυρίας Χάντζλικ ε, που μιλούν για απαγόρευση υψηλότερων διατραπεζικών ε, προμηθειών σε σχέση με αυτές που προβλέπει ο κανονισμός. Συμφωνώ, αλλά για λόγους ασφάλειας δικαίου πιστεύω ότι θα έπρεπε ίσως να το συμπεριλάβουμε στο άρθρο 5 και να μην χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Αν συμφωνεί η κυρία Χάντζλικ, ε, τότε ούτως να πράξουμε. Μία νέα προσέγγιση προτείνουν κάποιες τροπολογίες και δεν συμφωνώ με αυτές τις τροπολογίες. Να αναφερθώ στις τροπολογίες που αφορούν ε, το θέμα, για παράδειγμα, του ψηφιακού πορτοφολιού. 30, 31, 34, 41 και 46. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτές τις τροπολογίες ε, και μπορεί να με διορθώσει αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι ούτω ή άλλω οι πληρωμέ που αναφέρονται, οι υπηρεσίε πληρωμών, ούτω ή άλλω διέπονται από τον κανονισμό. Εδώ ο κανονισμό ε, διέπει την χρήση των καρτών και τι σχετικέ πληρωμέ, ανεξαρτήτω αν γίνεται μέσω ε, τηλεφώνου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δείτε για παράδειγμα το 7 ε, και 17 του άρθρου 2. Θα το δείτε. Το 7 καλύπτει τις συναλλαγές μέσω οποιοδήποτε μέσου που έχει σχέση με κάρτα, τηλεπικοινωνιών, ε, ε, άλλου λογισμικού κλπ. Το σημείο 17 μας λέει επίσης ε, ότι το μέσο πληρωμής που βασίζεται στην κάρτα μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Κάρτα, τηλέφωνο, υπολογιστής ή οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό μέσο με τις κατάλληλες εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο, εκείνος που πληρώνει για να καταβάλει την πληρωμή, για να κάνει τη συναλλαγή. Ο κανονισμός λοιπόν καλύπτει όλες τις διατραπεζικές προμήθειες και δεν εξαιρεί όσες ε, υπηρεσίες ε, χρησιμοποιούν την πραγματική κάρτα. Όσον αφορά το ψηφιακό ε, πορτοφόλι. Αν θέλετε να υπάρξουν επιπλέον ε, τρόποι πληρωμών ε, που θα συμπεριληφθούν, θα ήθελα να σας παραπέμψω στο 17 που μιλάει για όλες τις συναλλαγές πληρωμών, εκτός από τα εμβάσματα και τις χρεώσεις, γιατί αυτά καλύπτονται από την οδηγία 260 ε, του 2012 το, ο, στα, ο σταθμισμένος μέσος όρος ε, σε πολλές τροπολογίες, μεταξύ των οποίων ε, το 56 και το, μεταξύ των οποίων η 56 και 63, πρόκειται για τροπολογίες τις οποίες εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω, γιατί η, λόγω της μεθόδου που χρησιμοποιείται για το σταθμισμένο μέσο όρο των διατραπεζικών προμηθειών θα υπάρχει πρόβλημα με τον έλεγχο του ποσού αυτού και το κατά πόσο ένα μέγιστο όριο έχει ξεπεραστεί. Γιατί οι εταιρείε που θα έχουν ε, το, τις πληροφορίες, ε, γιατί τα, τα δεδομένα ε, αυτά πρέπει να είναι γνωστά προκειμένου να μπορούμε να υπολογίσουμε το σταθμισμένο μέσο όρο. Επίσης, οι τροπολογίες δεν συμπεριλαμβάνουν ενημέρωση, πληροφορίες σε σχέση με το ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Οι εταιρείε πληρωμών με χρήση καρτών Ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Η μέγιστο, ο μέγιστος σταθμισμένος μέσος όρος για τις διατραπεζικές προμήθειες θα σήμαινε ότι οι εταιρείε καρτών θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν, να επιβάλλουν διαφορετικά τέλη για διαφορετικές συναλλαγές, δηλαδή για διαφορετικά είδη καρτών ή για διαφορετικά είδη υπηρεσιών ή προϊόντων ε, ή ε, σε διαφορετικούς ε, τόπους τους οποίους έγιναν οι συναλλαγές. Οπότε θα υπάρχουν κάποια τέλη πάνω από το μεσόρο και κάποια τέλη κάτω από το μεσόρο που σκοπό θα έχουν ε, το, το ποσό, το συνολικό, ο μέσος όρος να είναι κάτω από το ε, κατώτατο όριο. Θα είναι δύσκολο επίσης να επιβάλλουμε κυρώσεις ε, αν ε, ο μέσος όρος αυτός ξεπερνιέται. γι αυτό, και σε αυτό στοχεύουν οι τροπολογίες αυτές. Νομίζω ότι ένας σταθμισμένο μέσο όρο ουσιαστικά θα αυξήσει τελικά το μέσο όρο των τελών. Και οι εταιρείε καρτών μπορεί να χρησιμοποιήσουν ε, τα τέλη δηλαδή στις ε, κανονικές πιστοτικές κάρτες να επιβάλλουν λιγότερα τέλη και πολύ ψηλότερα τέλη για premium κάρτες, για golden κάρτες και ούτω καθεξής. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους σε σχέση με τον όγκο συναλλαγών. Τώρα, τα κρυμμένα, οι κρυμμένες διατραπεζικές προμήθειες, 41, 42 και 71 τροπολογίες. Πάλι με δυσκολεύουν αυτές οι τροπολογίες. Το σημείο 22 λέει ότι τα τριμερή συστήματα όταν πρόκειται και για εκδότες και για αποδέκτες, θα πρέπει να θεωρούνται τέτραμερή συστήματα. Και ο κανονισμός το καλύπτει ήδη αυτό στις τροπολογίες, ωστόσο, προβλέπεται ξεχωριστή λογιστική για τους εκδότες και για τους αποδέκτες των, κρατών, των καρτών. Δηλαδή αντιμετωπίζει το θέμα αυτό σαν να είναι δύο διαφορετικά εντελώς θέματα, σαν να είναι δύο διαφορετικές, ε, ε, ε, σαν να είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Όμως δεν ισχύει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας κανονισμός μπορεί να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία μιας εταιρείας. Αν δει κανείς και το μερίδιο αγοράς αυτών των εταιριών είναι περίπου 1%. Πρόκειται λοιπόν για πολύ μικρό μερίδιο αγοράς και για αυτό το λόγο δεν βλέπω το λόγο τόσο σημαντικής παρέμβασης. Αν η κυρία Χάντλικ συμφωνεί, ε, θα μπορούσαμε θα μπορούσαμε να, να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό ε, με την ε, τροπολογία, λαμβάνοντα υπόψη και την τροπολογία της κυρίας Βερνιό, την υπαριθμό 91, και να δούμε την εξέλιξη τη αγορά μετά την εφαρμογή του κανονισμού, αν χρειάζεται ε, στη συνέχεια και θεωρηθεί απαραίτητο τα τετραμερή συστήματα να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Θα στείλω κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε του σκιώδη κατά τι επόμενε εβδομάδε. Θα ήθελα να οργανώσω μία συνάντηση με του σκιώδη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το χρονοδιάγραμμά μας μπορούμε στις 10 Φεβρουαρίου να εξετάσουμε τις συμβιβαστικέ και να τις ψηφίσουμε στις 11. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων θα ψηφίσει στις 20 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες, ευχαριστώ το προσωπικό και ευχαριστώ και όλους και όλους Ελπίζω να συνεχίσει η επικοδομητική μας ε, δουλειά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίλαν για αυτήν την ε, εκτενή παρουσίαση των θεμάτων και των επίμαχων. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα θα κοιτάξουμε να συζητήσουμε στις 10 για τις συμβιβαστικές πριν ψηφίσουμε στις 11. Τώρα, οι σκιώδεις θα μας πούν τα σχόλιά τους για τις τροπολογίες. Ο κύριος Μπορισόφα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες με διάφορες ιδέες για τα βασικά θέματα ε, με σκοπό να βρεθεί αποδεκτή συμβιβαστική λύση. Εφιστώ την προσοχή σας στα βασικά ε, τριμερή, τετραμερή συστήματα. Εδώ μόνο στα τετραμερή θα τα μειώσει, δεν θα καλύπτονται τριμερή, δεν δίνει λόγο. Ε, ο λόγος είναι η, το μικρό μερίδιο αγοράς. Έχουν δυσκολία οι διερμηνείς να σας παρακολουθούν. Ε, λίγο πιο αργά παρακαλώ. Ιδιαίτερα διαβάζετε κείμενο που δεν το έχουν οι διερμηνείς. Λοιπόν, για τις προμήθειες και τις εμπορικές τράπεζες και τα τριμερή συστήματα που δεν έχουν διαφάνεια έλεγα. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που ρυθμίζουν τις κάρτες όπως οι διατραπεζικές τα τραμερή συστήματα για να έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού χωρίς τρέβλωση. Εγώ δεν έβαλα τροπολογίες γιατί νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις ο ανταγωνισμός οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα μέσω και πρόθεσμα, δηλαδή χαμηλότερες προμήθειες. Όμως συμφωνώ με τις τροπολογίες που ρυθμίζει στα τριμερή συστήματα ε, την κατάσταση σύμφωνα με το ψήφισμα του 2012 του Νοεμβρίου του Κοινοβουλίου που λέμε ε, ότι τα μικτά, οι μικτές πληρωμές και τα τριμερή συστήματα μπορεί να ε, ε, τονώσουν τον ανταγωνισμό ναι, και θέλουμε ίσους κανόνες ανταγωνισμού για διαφάνεια. Επίσης και άλλες καινοτόμοι μορφές όπως ψηφιακές πρέπει να διατηρηθούν η ανάπτυξη της αγοράς ε, για τις ηλεκτρονικές ε, πληρωμές και μετακινητά αυξάνεται αλλά ακόμα είναι ευαίσθητη και περιορισμένη. Και ε, αν είμαστε πολύ υπαγορευτικοί θα δημιουργήσουμε εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επίσης αναφέρομαι πάλι στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Ε, τώρα άρθρα 3 και 4 για ανώτατα όρια στις ε, προμήθειες. Συμφωνώ με την πρόταση της ε, Κομισιόν να έχει ανώτατα όρια παντού. Είναι σημαντικό για, τη για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Είναι σημαντικό και για την κινητικότητα των πολιτών. Νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε οι περισσότεροι συνάδελφοι για το άρθρο 4 σχετικά με τις προμήθειες ε, για τις ε, συναλλαγές. Ε, εδώ διαφέρει η κατάσταση στα κράτη-μέλη και πρέπει να βρούμε μια λύση που θα εξυπηρετεί τους περισσότερους. Έχω προτείνει σταθμισμένο μέσο όρο που αντικατοπτρίζει τις διάφορες μορφές πληρωμών με κάρτες Φοβάμαι ότι όταν δεν είναι πολύ αναπτυγμένη η αγορά, τα ανώτατα όρια θα τα αυξήσει, όπως για τις εκδόσεις κρατών. Και τέλος, ο καταναλωτής θα υπομειστεί το κόστος. Επίσης υπάρχουν διάφορα προϊόντα, ε, συναλλαγές υψηλού και χαμηλού κόστους, είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε ούτως ώστε να ε, γίνονται οι πληρωμές. Άλλα θέματα ελέγχου. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να συσκεφτούμε περισσότερο το σύστημα. Η Κομισιόν τα προηγούμενα δέκα χρόνια είχε ρυθμίσει το μέσο κόστος. Υπάρχουν τροπολογίες υπέρ της λύσης αυτού του θέματος. Σύμφωνο και με τις τροπολογίες για τον ορισμό των πληρωμών με κάρτες. Δεν πρέπει να παρακάμπτεται το άρθρο 24 επίσης. Θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι όταν χρησιμοποιούν τις κάρτες οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν τις διάφορες δυνατότητες λειτουργίας για να μην παραπλανώνται. Θα συνεχίσουμε με τους σκιώδεις να αναζητούμε κατάλληλες λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που μας τα είπατε τόσο καθαρά. Η κυρία Βερνιό. Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως σας είπα και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει ως στόχο να βάλει λίγη τάξη σε όλο αυτό το θολό τοπίο που έχουμε όσον αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα μιλήσει και στο παρελθόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα αυτό όσον αφορά τις ε, πληρωμές αυτές όταν είχαμε συζητήσει για τα εμβάσματα, τα αυτόματα εμβάσματα. Δεν είχε ενδιαφερθεί τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των καρτών. Να ευχαριστήσω πάντως τον εισηγητή τον κύριο Μπιελάν για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή και είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στην ομάδα εργασίας των σκιωδών στο Στρασβούργο. Συμφωνώ με τη δική σας την άποψη ότι θα έχουμε σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όσον αφορά το σταθμισμένο μέσο όρο. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό ζήτημα, ένα δύσκολο ζήτημα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει περαιτέρω να καταστήσουμε το σύστημα πιο πολύπλοκο. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες μου. Όντως η 60, η τροπολογία 60 προτείνει μια αύξηση στο 0,3% όσον αφορά τις προμήθειες. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να προτείνουμε ένα ανώτατο όρο για τις προμήθειες αυτές. Είναι πολύ υπερβολικές σε κάποιες χώρες και νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε μία μικρή αύξηση προκειμένου τα κράτη-μέλη να έχουν υψηλότερο βαθμό ευελιξίας και να καταφέρουν τελικά να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς, καθώς επίσης και στα όσα ισχύουν για το τραπεζικό τομέα σε κάθε χώρα, Θέλοντα παράλληλα λοιπόν ένα ανώτατο όρο το οποίο γενικά είναι αποδεκτό. Αναφέρομαι κυρίω στι τράπεζε εκείνε, οι οποίε δεν εξυπηρετούν πάρα πολλού εμπόρου, αλλά έχουν πολλού πελάτες με ένα χαμηλό οικονομικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα τα ταμιευτήρια. Θεωρώ λοιπόν ότι το 0,3% θα πρέπει να είναι ένα ανώτατο όριο και βέβαια κάθε κράτος μέλος μπορεί να θέσει και χαμηλότερο όριο. Το ο στόχος είναι να μειώσουμε τις προμήθειες για τους εμπόρους, προκειμένου να μπορούν ενδεχομένω να μειώσουν και τις τιμές τους, πραγματοποιείται δεδομένο, τότε η μείωση αυτών των διατραπεζικών προμηθειών θα πρέπει όντως να γίνεται, να καταγράφεται ουσιαστικά από τους αποδέκτες, από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας και στη συνέχεια να μετακυλείεται το αυτή η μείωση του κόστους και στους πελάτες. Στη συνέχεια έχουμε και το σύστημα το τριμερές, το οποίο τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλησε να εντάξει στην έκθεσή της. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ένα σύστημα όπου έχουμε διατραπεζικές προμήθειες κρυφές και ιδιαίτερα υψηλέ. Και σε ορισμένε χώρε υπάρχουν κάποιοι έμποροι οι οποίοι δεν δέχονται συγκεκριμένε κάρτε, συγκεκριμένα μέσα πληρωμή, ακριβώ επειδή υπάρχουν αυτέ οι υψηλέ κρυφέ προμήθειε. Ξέρετε ότι οι κάρτες αυτές στις οποίες αναφέρομαι έχουν να κάνουν με ένα συγκεκριμένο προφίλ πελατών, με ένα συγκεκριμένο προφίλ καταναλωτών και νομίζω ότι μέσω της τροπολογίας μου αυτή προσπάθησα να προσδώσω ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας. Σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι με την τροπολογία 91. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί επισταμένως με το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Μπιλάν και ελπίζω θα καταφέρουμε να καταλήξουμε συμφωνία και με εσά και με τις υπόλοιπε πολιτικές ομάδες την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς θα μιλήσει για τον κύριο Σμιτ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα συζητήσω τις τροπολογίες γιατί δεν τις ξέρω. Εγώ έχω ένα σημείωμα του κυρίου Σμιτ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στις προ... προμήθειες υπάρχει ένα ποσοστό αλλά δεν ικανοποιούνται οι καταναλωτές γιατί πρέπει να πληρώνει κανείς ε, κάθε ώρα όταν είναι σύμβουλος και αυτό μπλοκάρει ε, την ε, όλη διαδικασία δανειοληψίας και υποθηκών. Ευχαριστεί τον κύριο Μπίλαν, ο κύριο Σμιτ. Δεν είναι πεπισμένος ότι χρειάζεται νομοθεσία για να αντιμετωπίσει ψηλές προμήθειες. Ως φιλελεύθερος θέλει η αγορά να τα ρυθμίζει αυτά τις ρυθμίσεις τιμών, αλλά επειδή η αγορά δεν το κατάφερε, απέτυχε δηλαδή, ε, θα ταχθεί υπέρ της πρότασης της Κομισιόν. Για το ανώτατο όριο, όλε Σμιτ συμφωνεί με, την με τον εισηγητή ότι οι εμπορικές κάρτες δεν πρέπει να εξαιρούνται. Ε, δεν υπάρχουν τεχνικοί οικονομικοί λόγοι για να αντιμετωπιστούν διαφορετικά αυτές οι κάρτες. Ο κύριος Σμιτ δεν είναι υπέρ να συμπεριληφθούν ε, τα ψηφιακά μέσα σε αυτή την οδηγία. Αν συμπεριληφθούν ε, μπορεί και τράπεζες να βρουν διαφορετικές λύσεις. Θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο για τα τέλη από τις κάρτες και αλλού να ρυθμιστούν άλλες τεχνικές πληρωμών. Τέλος, ο Όλε Σμιτ δεν είναι υπέρ του σταθμισμένου μέσου όρου. Μπορεί να χρειάζεται ευελιξία, αλλά η διαφοροποίηση μεταξύ τομέων θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου θα είναι λιγότερη η διαφάνεια και η κατανόηση των αγορών πληρωμών. Και αυτό είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε, συμπεραίνει. Και τέλος ευχαριστεί τους πάντες και προσβλέπει στην επόμενη συνεδρία των σκιωδών. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και τον εισηγητή και, τις, και τους Η κυρία Χάνσλικ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή ως σκιώδης. Έκανε πάρα πολύ δουλειά στο φάκελο αυτό. Συμφωνώ με τον εισηγητή τις τροπολογίες μου για το άρθρο και 4 να τις πάω στο άρθρο 5. Καλή ιδέα ακούγεται αυτή πόσο μάλλον που ε, εγώ και ο προηγούμενος ομιλητής απορρίπτουμε 100% την ιδέα του σταθμισμένου μέσου όρου, που είναι τελείως ασαφής για τους εμπόρους από ό,τι φαίνεται. Εμείς θέλουμε διαφάνεια, καθαρότητα στο κάτω-κάτω. Αν εισαγάγουμε σταθμισμένο μέσο όρο θα τα χάσουμε αυτά. Όσο λιγότερη σύγχυση δημιουργηθεί τόσο το καλύτερο και πρέπει να το σκεφτούμε πολύ πριν πιάσουμε σταθμισμένο μέσον όρο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στα κάτωθη. Ο αντίκτυπος των διατραπεζικών προμηθειών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις δεν μπορούμε να επιδεινωθεί για τις ΜΜΕ η κατάσταση. Δεν μπορεί να μειώσουμε τις διατραπεζικές προμήθειε ωφελώντα κάποιους μόνο στην αγορά, κάποιε οντότητε που είναι ήδη σε θέση ισχύω. Τράπεζες εννοώ. Και τους παρόχους υπηρεσιών ενώ κατά τον ίδιο χρόνο οι τράπεζες θα σταθμίσουν τα χρήματα που έχασαν από τους μεγάλους χρεώνοντας περισσότερο τις ΜΜΕ που είναι μικρότερες οντότητες στην αγορά. Πρέπει να προσέξουμε πολύ αυτό το θέμα, τον αντίκτυπο που θα έχουν όλα αυτά στις ΜΜΕ. Ζητώ λοιπόν από τον εισηγητή να σκεφτεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Τώρα, η Κομισιόν να μας πει. Η κυρία Βίζενμπεκ πρώτη, νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον εισηγητή για το ότι κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα να επιτελέσει ένα πάρα πολύ θετικό έργο και να ευχαριστήσουμε γενικότερα και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για όλες αυτέ τις τροπολογίες που καταδεικνύουν πραγματικά ότι γνωρίζετε πολύ καλά πώ λειτουργεί εν λόγω αγορά και εν γέννη δείχνετε μια επικοδομητική προσέγγιση. Σα ευχαριστούμε λοιπόν. α περάσουμε τώρα πρώτα στα σχόλια του εισηγητή. Και εμεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνούμε με τον εισηγητή όσον αφορά την αξιολόγηση των τροπολογιών που έχει κάνει για κάποια λεπτομερή ζητήματα, για το αν θα πρέπει δηλαδή να αναφέρουμε τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν χαμηλότερες προμήθειες, νομίζουμε ότι καλύπτεται αυτή η δυνατότητα, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνεται μας τροπολογίας. Επίσης, η απαγόρευση υψηλότερων προμηθειών υφίσταται, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνεται στο κείμενο αυτό. Εσείς βέβαια θα αποφασίσετε για το αν θα διατηρήσετε τη διάταξη αυτή ή όχι. Τώρα, όσον αφορά το ηλεκτρονικό ψηφιακό πορτοφόλι, πολύ. Ο συνάδελφό μου εδώ πέρα μπορεί να σα δείξει το δικό του το πορτοφόλι, ουσιαστικά για να καταλάβετε τι είναι αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι. Είναι η ηλεκτρονική εκδοχή αυτού του πράγματο που κρατάω στο χέρι μου. Ουσιαστικά. Ναι. Θεωρούμε λοιπόν και εμεί ότι δεν είναι αναγκαίο να αναφερθούμε συγκεκριμένα στο ψηφιακό πορτοφόλι αναφερόμενοι σε όλες τις δυνατότητες πληρωμής, σε όλες τις ηλεκτρονικές δυνατότητες πληρωμής, καλύπτουμε και το ψηφιακό πορτοφόλι. Νομίζουμε ότι θα δημιουργήσει σύγχυση το να αναφέρουμε το ψηφιακό πορτοφόλι ως ξεχωριστή αυτόνομη πληρωμή, γιατί δεν είναι στην ουσία. Όσον αφορά το σταθμισμένο μέσο όρο, πολλοί σκιώδεις ηγητής αναφέρθηκαν σε αυτό. Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μην προχωρήσει σε σταθμισμένο μέσο όρο, αλλά σε ένα απόλυτο ανώτατο όριο. Και γνωρίζουμε ότι ο σταθμισμένος μέσος όρος πολλές φορές έχει γίνει αποδεκτός και αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ιδίως όταν συζητούσαμε τα δύο διεθνή αυτά συστήματα, τα οποία δεν θέλανε να αποδεχθούν κανένα απολύτως όριο. Τα δύο αυτά λοιπόν συστήματα μας ζητούσαν μια κάποια ευελιξία όσον αφορά το μέσο όρο, προκειμένου να μπορούν να προσαρμόσουν και τις προμήθειές τους. Στα πλαίσια της συνένεσης ενός εμβιβασμού ουσιαστικά είχαμε αποδεχθεί τότε τον σταθμισμένο αυτό μέσο όρο. Είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε να αναλύαμε περισσότερο τις προμήθειες, να δούμε πώς εφαρμόζονται σε κάθε σύστημα. Η όλη όμως αυτή η εργασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, χρειάστηκε να αναλώσουμε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποίησαμε την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν συγκεκριμένες εταιρείες συμβούλων, ιδίως όσον αφορά τη χρήση Mastercard και Visa, και αν θέλουμε ουσιαστικά να καταλήξουμε με ομοιόμορφες προμήθειες, πρέπει πρώτα να δούμε αν ο σταθμισμένος μέσος όρος μπορεί να ισχύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ισχύει ένα χώρα, ανα τράπεζα, πώς ακριβώς θα διευθετηθεί. Και δεν ξέρω επίσης και αν τα κράτη-μέλη θέλουν πραγματικά να αφιερώσουν πολύ χρόνο μέσω των δικών τους εθνικών αρχών για να ασχοληθούν με το ζήτημα των σταθμισμένων μέσων όρων. Θεωρούμε ότι τα ανώτατα όρια αποτελούν μια καλύτερη λύση γιατί επιτρέπουν τελικά στους εμπόρους να δουν τελικά αν οι κανόνες λειτουργούν στην πράξη. Αν έχουμε σταθμισμένο μέσο όρο, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάει ένας έμπορος σε μια τράπεζα να παραπονεθεί για τις διατραπεζικές προμήθειες και η τράπεζα να του πει ότι κινούμεθε σε ένα σύστημα σταθμισμένων μέσων όρων και ότι επιτρέπω ότι σε αυτές, υψηλότερε ή, ή χαμηλότερες προμήθειες. Όσον αφορά τώρα τα τριμερή συστήματα. Όταν καταρτίζαμε την πρόταση αυτή, θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Είναι λογικό λοιπόν να μα ζητάτε τη συμπερίληψη των τριμερών συστημάτων. Έχουμε εντοπίσει όμω δύο σχετικά προβλήματα. Πρώτον, τα τριμερή αυτά συστήματα έχουν περιορισμένο μερίδιο τη αγορά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, κανένας ε, λιανέμπορος ε, δεν θα βρεθεί εκτό αγορά αν απορρίψει τελικά την πληρωμή με American Express. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεύτερον τώρα, το δεύτερο πρόβλημα που είχαμε εντοπίσει δεν ξέρουμε πώς είναι δυνατόν από νομικής πλευράς στα πλαίσια μιας εταιρείας να δούμε ακριβώς πώς περνάμε από τη μία προμήθεια στην άλλη, ποια είναι η όλη αλυσίδα τελών και προμηθειών. Για αυτό το λόγο αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να ρυθμίζουμε τα συστήματα αυτά μόνο όταν χρησιμοποιούν τράπεζες αδειοδότησης και ουσιαστικά Θέλουμε όταν έχουμε τριμερή συστήματα να προβλέπουμε τη δυνατότητα απόρριψης μιας κάρτας αν οι προμήθειες είναι πολύ ψηλές και να μπορούν ουσιαστικά οι έμποροι ή οι καταναλωτές να κάνουν την σωστή για αυτούς επιλογή αν οι καταναλωτές επιθυμούν να πληρώσουν ένα υψηλότερο τέλος για να χρησιμοποιήσουν American Express και να έχουν όμως όλα τα υπόλοιπα ωφέλη τα οποία μπορεί να αποφέρει η κάρτα αυτή, όπως για παράδειγμα μίλια ή ούτω καθεξής, τότε θα αποφασίσουν μόνοι τους ότι θα κάνουν κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά θέλουμε μια συνειδητή επιλογή εμπόρων και καταναλωτών. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι πετυχαίνουμε και την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα τα οποία υφίστανται στην αγορά. Άλλα ζητήματα τώρα. Συζητήσαμε το σταθμισμένο μεσόρο. Ας περάσουμε τώρα σε κάποιο άλλο ζήτημα. Αν θα πρέπει να ρυθμίσουμε και τα τέλη εκείνη τα οποία επιβάλλονται από την εμπορική τράπεζα στον έμπορο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε εδώ πέρα ότι όντως τα προνόμια τα οποία περνάνε από τον ένα φορέα στον άλλον. Αν υπάρχει ένας σημαντικός ανταγωνισμός από την πλευρά των αποδεκτών, τότε οι τράπεζες μετακυλίουν τα πλονεκτήματα που έχουν από τα χαμηλότερα τέλη, από τις χαμηλότερες προμήθειες και τη διαφορετική περίπτωση οι έμποροι θα απευθυνθούν σε κάποια άλλη τράπεζα. Έτσι λοιπόν όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω μιας άλλης οδηγίας, της οδηγίας για τις πληρωμές, είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας, είχε προβλέψει τότε τη δυνατότητα αυτή. Σε επίπεδο τώρα αποδέκτη, νομίζουμε ότι ο ανταγωνισμός αυτός μπορεί να λειτουργήσει. Αποφασίσαμε λοιπόν να μην ρυθμίσουμε τα τέλη αυτά, τα market service charges. Νομίζω ότι έχω καλύψει όλα τα σημεία στα οποία ήθελα να αναφερθώ. Να δώσω το λόγο τώρα στον αδελφό μου. Ένα θέμα μόνο να θέσω, το επίπεδο των ορίων, ε, την πιθανή αύξηση για να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο για τα κράτη-μέλη να ε, τα μειώσουν με τη σειρά τους. Κατά την άποψή μας, το επίπεδο των ορίων ε, μπορεί να είναι 0,2-0,3%. Ε, Visa, Mastercard και ε, την ομάδα των, των τραπεζικών καρτών της Γαλλίας, τον όμιλο τραπεζικών καρτών της Γαλλίας αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τα νούμερα αυτά είναι να εξασφαλίσουμε ότι ένα μερίδιο του ωφέλου της χρήση των καρτών ε, να μετακυλίεται στους εμπόρους και στους καταναλωτές. Και πιστεύουμε ότι το 0,2 και 0,3 το κάνει αυτό ενώ τα παραπάνω επίπεδα ε, δεν, θα, ε, δεν θα σημαίνουν ότι θα μετακυλιστεί το όφελος στους καταναλωτές και τους εμπόρους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Νομίζω ότι ήταν πολύ λεπτομερής και επικοδομητική η συζήτηση. Να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Μπίλαν, εκτός αν θέλει κανένα άλλο συνάδελφος ε, να θέσει ερωτήματα προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Ωραία, τότε ο κύριος Μπίλαν, για να συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Βερνιό, ε, Χάντλικ, ε, ε, Μάντερ, το εκ του κυρίου Σμιτ, που υπέβαλαν τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή για την εξαιρετική συμβολή της στη συζήτηση. Νομίζω ότι διασκέδασαν κάποιες αμφιβολίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω, όπως είπα, να συντάξω τις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, κατά τις επόμενες εβδομάδες. Δεν θα καλύψω όλες τις τροπολογίες βέβαια, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να συμπεριλάβω στο δυνατόν περισσότερες. Θα προσπαθήσω να οργανώσω συνάντηση σκιωδών την εβδομάδα του Στρασβούργου. Μία ακόμη φορά ευχαριστώ πάρα πολύ το προσωπικό της Επιτροπής γιατί με βοήθησε στην προετοιμασία της νομοδότησης αυτής. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ολοκληρώνονται οι εργασίες μας ε, για σήμερα. 10 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Θα έχουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη για να συζητήσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και όπως λέμε θα ψηφίζουμε την 3η 11 Φεβρουαρίου, συνήθως το πρωί και το απόγευμα θα έχουμε άλλη μία συνεδρίαση ε, το απόγευμα της 11ης ε, Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας, τη σημαντική δουλειά σας για το θέμα αυτό, όπως επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έσπευσε να έρθει Βλέπετε ότι άξιζε πάρα πολύ τον κόπο. Ε, εμάς μας ικανοποίησε όλος ιδιαίτερος που ακούσαμε τη δική σας συμφωλή. Ευχαριστώ να ξανακούσουμε τις απόψει, σα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα, γιατί ακούμε, λαμβάνουμε διαφορετικά μηνύματα από διαφορετικούς ανθρώπους και είναι καλό να υπάρχει σαφήνεια γύρω από τη συζήτηση και επαφίεμαι στον κύριο Μπίλαν και τους κοιόδης συζητητέ να καταλήξουν σε μια εξισορροπημένη ε, πρόταση που θα ωφελήσει και του επιχειρηματίε αλλά και του καταναλωτέ. Αν δεν σας δω την επόμενη εβδομάδα ε, στο Στρασβούργο, θα τα ξαναπούμε στις 10 Φεβρουαρίου.